Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχουμε την πιο εντατική και σίγουρα την πιο εκτενή συνεδρίασή μας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να, αποταθούμε, να αποφαθούμε σχέση ε, με 1902 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί επί του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2016. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Εισηγητή και, το, και εισηγητή για τα λοιπά τμήματα για το έργο τους που χαρακτηρίστηκε από μεγάλη επιμέλεια και καταπώνητη εργασία. Νυχθημερών προσπάθησαν και εργάστηκαν και οι εισηγητέ και η γραμματεία και τους ευχαριστώ όλους θερμά για την συνεργασία τους προκειμένου να δημιουργήσουμε τι καλύτερες προϋποθέσεις για την ψηφοφορία αυτή του προπολογισμού. Βέβαια υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες και το να προβλέψουμε τι θα συμβεί το 2016 είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και δεν αποκλείεται στο εγγύ μέλλον να, χρειαστεί να τροποποιήσουμε τον προπολογισμό μας. Πολλά δε μάλλον που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνέλθει, θα συνεδριάσει την Τετάρτη το πρωί για να εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2015. Κάτι που θα επηρεάσει και τον προϋπολογισμό του 2006 σε ό,τι αφορά και τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές. Η κυρία Γεωργίευα, η αρμόδια επίτροπος για τα δημοσιονομικά θέματα, θα έρθει αμέσως μετά την συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το μεσημέρι το απόγευμα της Τετάρτης. Οπότε ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει τις ψηφοφορίες μέχρι τότε και να οργανώσουμε και μια επιπλέον συνεδρίαση για την ακρόαση με την Επίτροπο Γεωργίευα. Είχαμε σκεφτεί αρχικά να γίνει τη Δευτέρα το απόγευμα στο Στρασβούργο. Κολλείεται όμως ε, για την ημερομηνία αυτή η κυρία Γεώργιεβα και πρότεινε να έρθει αμέσως μετά τη συνεδρίαση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας ενημερώσει. Το Συμβούλιο θα αποφανθεί στις 21 Οκτωβρίου και κατόπιν θα επιληφθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του πακέτο της μετανάστευσης. Επίσης και έπρεπε αυτό να είχα ξεκινήσει. Θα ήθελα πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Κυρία Γορδιασάβαλ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν τροπολογίες για τον υπερθμό 6 διορθωτικό προπολογισμό, θα ήθελα να το συμπεριλάβουμε στην αυριανή μας ψηφοφορία μετά την ψηφοφορία του Γενικού Προπολογισμού, γιατί δεν μπήκε αυτεπάγγελτα στην ημερήσια διάταξη, γιατί είχε ήδη εγκριθεί και αποστάλει. Αλλά μια και δεν υπάρχουν τροπολογίε και δεν υπάρχουν και προβλήματα, θα μπορούσαμε κάλλιστα να ψηφίσουμε αύριο για το θέμα αυτό. Ε, αύριο ή μεθαύριο, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Οπότε η έκθεσή σας θα ακολουθήσει την ψηφοφορία του προπολογισμού του 2016, μια και δεν υπάρχουν και τροπολογίες. Ωραία. Τροποποίησαμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη και να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις των συντονιστών στη συνεδρίαση της 15 Σεπτεμβρίου και στη σημερινή συνεδρίαση. Καταρχήν, ζητήσαμε από τη διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών την άδεια να εκπονήσουμε έκθεση πρωτοβουλίας με θέμα το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, ζητήσαμε κατά εφαρμογή του άρθρου 54 ε, την άδεια να συντάξουμε γνωμοδότηση επί της εκθέσεως της Επιτροπής Απασχόλησης με θέμα την έκθεση εφαρμογή ε, για τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην περίοδο 2007-2014. Αποφασίσαμε επίσης να συντάξουμε γνωμοδότηση για τις διαδικασίες προκειμένου ε, να γίνουν εφικτοί το ΦΠΑ και το ΑΕΜ με βάση τις ε, προτάσεις και τα μέτρα για να, ε, ε συντρέξουν οι προϋποθέσεις πληρωμής. Ο κύριος Λεβαντόφσκι είναι ο εισηγητής και επίσης η Ιζαμπέλ Τομά είναι αρμόδια για τον αθεώρηση του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου μαζί με τον Γιάννο Ολμπρίχτ. Ζητήσαμε και την εκπόνηση δύο μελετών τη μελέτη για την αναθεώρηση του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου. Σας είπα ποιοι θα είναι οι δύο συνεισηγητές για το θέμα αυτό. Και επίσης ζητήσαμε και συγκριτική μελέτη για το κόστος ε, του κάθε ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι ευρωπαϊκές πολιτικές στα κράτη-μέλη δεν ορίστηκε ακόμη συγκητής για το θέμα αυτό. Επίσης, συμφωνήσαμε να στείλουμε επιστολή επισημένοντας τα, προβλήματα που έχουμε με το χρονοδιάγραμμα και τη συμβατότητά του με τη ε, διαδικασία του περιπολογισμού. Κατά την ψηφοφορία, την εξέταση και την συνδιαλλαγή για τον επόμενο προϋπολογισμό, δηλαδή του 2017. Επίσης, ε, ο Ευρωπαίος Διαμοσολαβητής ε, μας υπέβαλε αίτημα να παραστεί στον τριμερή διάλογο. Και μια και έστειλε το ίδιο αίτημα στις επιτροπές ΑΦΚΟ, ΚΟΝΤ και ΛΥΜΠΕ, εκτός από τη δικιά μας, σκέφτηκα, σκέφτηκα με τους συντονιστές ότι καλό θα ήταν να συνεννοηθούμε και με τις υπόλοιπες επιτροπές για να υιοθετήσουμε μια ενιαία προσέγγιση. Επίσης, προτείναμε και αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε τους ευρωβουλευτές που είναι μέλη της ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους σπόρους να προσέλθουν στην Επιτροπή μας μέχρι τα τέλη του έτους. Επίσης, συμφωνήσαμε να κρίνουμε το αίτημα των Startups Europe των μαθητών ε, μεγάλων, των, των Grand Ecole και των ε, σχολών ε, διαχείρισης της Γαλλίας να έρθουν να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα της Ολομέλειας για το σεμινάριό τους. Και επίσης έχουμε και κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών με θέμα τις προκλήσεις που ανακύπτουν για τον προϋπολογισμό εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών και της κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία. Όσοι συμμετείχαμε τον περασμένο Ιούλιο στην αποστολή στη Σικελία, να κάνουμε μια ενημέρωση για τα αποτελέσματα αυτής της αποστολής προς συναδέλφους. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μου. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην εξέταση των τροπολογιών και στην ψηφοφορία του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2016. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να βεβαιωθώ ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης 3η Σεπτεμβρίου που σας έχουν διανεμηθεί σας βρίσκουν σύμφωνος. Δεν βλέπω να ζητά κανείς ε, το λόγο για τα πρακτικά, οπότε θεωρώ ότι εγκρίνονται. Και τώρα ο λόγος στους ηγετές μας για να μας κάνουν μια εισαγωγή για την εξέταση των τροπολογιών και την ψηφοφορία. Πρώτα ο κύριος Φερνάντες, που είναι ο Γενικός Συγητής για το προπολογισμό του 2016. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες και όλους τους κοιόδους συγητές, όλους τους συντονιστές για το έργο τους που ξεκίνησε με δύο ψηφίσματα. Στις αρχές του έτους ήταν το πρώτο και τον Ιούλιο το δεύτερο, στο οποίο αποφασαφινίστηκε η εντολή της διαπραγμάτευσης. Με προτεραιότητά μας να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε να συνδράμουμε τους πρόσφυγες και να λύσουμε το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Και επίση ε, τα τρία βασικά θέματα ήταν η απασχόληση, οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά ήταν οι στόχοι του προπολογισμού για το 2016, πρωταρχική. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για τη βοήθειά τους, ε, ε, γιατί έτσι καταλήξαμε σε ένα έγγραφο στο οποίο δείχνουμε τη συσπήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί όλοι στηρίζουμε αυτούς τους στόχους. 1902 τροπολογίες έχουν κατατεθεί, κάτι που δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον ε, και την προσήλωση των συναδέλφων σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και θα έχουμε μια αρκετά εκτενή συνεδρίαση σήμερα προκειμένου να ψηφίσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Πάντως σας ευχαριστώ θερμά γιατί καταλήξαμε σε μια σύμπνοια μεταξύ των πολιτικών ομάδων και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη γραμματεία και όλους ιδιαίτερους τον Κιγιόμ που κάθεται εκ δεξιών για την ακαταπώνητη προσπάθειά του και επίσης να ευχαριστήσω και τους συμβούλους των πολιτικών ομάδων και κυρίως τις συμβούλους με τους οποίους είχαμε στενή συνεργασία από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά να ευχαριστήσω τους ε, συμβούλους και όλων των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων, γιατί όλοι συνέβαλαν στο να καταλήξουμε σε αυτό το ποιοτικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, χρειάστηκε μια ολόκληρη Κυριακή να αφιερώσουμε την ε, γραμματεία στην εξέταση όλων των γραμμών των προπολογισμού και των τροπολογιών και θα ήθελα να επενέσω τη Γραμματεία για την ε, αξιέπαινη προσπάθειά της, αλλά ταυτόχρονα και τις πολιτικές ομάδες και τους συμβούλους, γιατί είναι πολλές φορές ε, αφανές αυτό το έργο, αλλά υπαρκτό και σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για την προσήλωσή σας, την επιμέλειά σας, ε, τη ζέση και την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γενική Εισηγητά. Εσείς ήσασταν συντονιστής ε, αυτού του του έργου, οπότε δεν μπορούμε παρά να συγχαρούμε και να ευχαριστούμε τον κύριο Ντεπρέ που είναι ο συντάκτης για τα άλλα τμήματα του προπολογισμού. Ο κύριος Ντεπρέ θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε, γιατί θα προτιμούσα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή πριν την ψηφοφορία για τα υπόλοιπα τμήματα, ούτως ώστε να μην ε, ε, διακόψω τη συγκέντρωσή σας μετά από την ε, πάρη μας κύριο Φερνάντες. Πρόεδρος. Βλέπω ότι είναι συναισθηματικά φορτισμένες οι, οι ώρες. Κύριε Καλβίνιο, τι λέτε. Μια που είναι τόσο ιδιαίτερες συνθήκε. θεωρείτε ότι μπορείτε ευθύ αμέσω να προβείτε σε μια δήλωση πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία. Καλβίνιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω για να είμαι σύντομη. Και επίσης θα προσπαθήσω να συγκρατήσω τα συναισθήματα που μας ξεχυλίζουν στα αγγλικά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριε Βουλευτέ τη Επιτροπή Προπολογισμού, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία μου δίνετε για να μιλήσω σε εσά πριν τόσο σημαντική ψηφορία, την οποία πρόκειται να διεξαγάγεται στι προηγούμενε συναντήσει, σε τριμερεί ε, συναντήσει και σε όλε τι επαφέ που είχαμε μπορέσαμε να σας παρουσιάσουμε το σχέδιο προπολογισμού για την χρήση του 16 και επίσης σα εξηγήσαμε ε, τι πρεσβεύουμε όσον αφορά ε, τη γνώμη του Συμβουλίου. Αλλά σήμερα θα ήθελα να σε επιστρέψω την προσοχή στι διάφορες εξελίξεις που έλαβαν χώρα από τότε που προτείναμε το σχέδιο προπολογισμού τον Μάιο. Και επίσης ε, για αυτά τα γεγονότα τα οποία επισήμανε και ο Πρόεδρος. Από τα τέλη Μαΐου, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε το σχέδιο προπολογισμού για το 2016. Είχαμε διάφορες εξελίξεις σημαντικές, οι οποίες έλαβαν χώρα και οι οποίες ε, απίτησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί, να επιδείξει υπευθυνότητα αλλά και ελεγγύη. Όμως τα γεγονότα περνούν τόσο γρήγορα και ίσως ε, έχουμε λησμονήσει. Πάντως το πρώτο σημαντικό γεγονός το οποίο έγινε τους τελευταίους μήνες ήταν η κρίση της Ελλάδας και στο πλαίσιο των μέτρων για βοηθήσουμε δηλαδή, αυτέ τι δύσκολε ώρε, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια αύξηση τη προχρηματοδότηση για τα διευθυντικά ταμεία. Για το πρόγραμμα 2014-2016 ε, και επίσης να υπάρξει και αύξηση του ρυθμού ε, δαπανών και το 5% που απέμεινε να εκταμεθεί πιο γρήγορα για τα προγράμματα του 2013. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα δις ε, για τον προηγούμενο του 2015. Αυτό κάτι τη γνώμη μας μπορούσε να καλυφθεί από τις πιστώσεις πληρών που είχαν εγκριθεί. Και, και το τονίζω, γιατί είναι σημαντικό για εσάς, χωρίς, λέγω, χωρίς να υπονομεύσουμε το στόχο του να μειώσουμε κατά 20 εκατομμύρια ε, αυτό το, το, το, το, τα πλήρωτα τα μάλλον για την ιδιωτική πολιτική επίση ε, για το 2016 και εδώ νομίζουμε ότι μπορεί να καλυφθούν αυτά τα οποία θέλουμε στα πλαίσια του σχεδίου προπολογισμού όπως προτείναμε. Τέλος πάντων θα σας ενημερώσω ενδελεχώς για το τι γίνεται όσον αφορά τις πληρωμές. Ακριβώς όπως έχει συμφωνηθεί. Η δεύτερη συναντησή μας θα είναι 19 Οκτωβρίου. Αμέσως μετά τις θερινές διακοπές είχαμε την κρίση για το γλακτοκομικό τομέα που και σε αυτή την περίπτωση ήταν ε, γεγονός που και αυτό έχει επίπτωση στον προπολογισμό. Ανακοινώσαμε μια δέσμη μέτρων για τα γαλακτοκομικά επίσης και την παροχή γαλακτός στους ε, πρόσφυγες. Αυτό στα πλαίσια των 500 ε, εκατομμυρίων δεν έγινε αντιληπτό. Εμείς όμως προσπαθήσαμε το κάθε ευρώ να χρησιμοποιηθεί για δύο σκοπούς. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί το γάλα για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών που ε, είχαν ανάγκη. Επίσης είχαμε τη δεύτερη τροπολογία το μέσα Οκτωβρίου. Επίσης είπαμε για κάποια μέτρα για προεκυπευτικά κατόπιν της παράτασης ε, του ρωσικού εμπάργου. Οπότε ε, ενημερώσαμε και τις προβλέψεις για τον γεωργοτομέα. Βεβαίω και η κρίση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για μακροχρονικό διάστημα. Είναι, πρόκειται για την κρίση που αφορά τους πρόσφυγες. Είναι κάτι χωρίς προηγούμενο. οπότε και τώρα έχουμε και πίεση χωρίς προηγούμενο επί του προϋπολογισμού μας. Το Κοινοβούλιο είχε δίκιο, γιατί στις καθημερινές γραμμές αυτό το είχε επισημάνει, το είχε θεωρήσει υψίστη προτεραιότητα και τότε είχε πει το Κοινοβούλιο ότι θα έπρεπε στο τίτλο 3 να το προβλέψουμε. Στο κονδύλιο μόνο 3, heading στα αγγλικά. Οπότε ήδη είχαμε 273 εκατομμύρια για δεσμεύσει περισσότερε πέραν των είχαμε προγραμματίσει για την κατανάστευση. Όμω χρειάζονται και άλλα μέτρα ούτω ώστε να καλύψουμε την ε, κρίση των προσφύγων. Ε, Επίση, ε, είχαμε και διάφορα άλλα πακέτα μέτρων και το τελευταίο ήταν την περασμένη εβδομάδα. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε την επανεγκατάσταση αυτών που χρειάζονται διεθνή προστασία, όπως συνεφώνησε το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Επίσης, οι επιπτώσεις θα αφορούν την ε, τροποποιητική επιστολή παριθμών 2 για το 2016. Είχαμε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, οπότε είπαμε για τον προορισμό του 2016 ποιες θα είναι οι επιπτώσει. 780 εκατομμύρια για αυτήν την μετεγκατάσταση ή επανεγκατάσταση, 600 για την χρηματοδότηση του ασύλου, ε, εσωτερική ασφάλεια και για την Frontex αλλά την EASO και την Europol. Και επίσης είπαμε να υπάρξει αναβάθμιση του εξωτερική δράση με την ανθρωπιστική βοήθεια. Είχαμε κάποιες δροπολογίε ε, δικέ σα. Ήδη καλύπτεται τους πόρους που χρειάζονται για αυτή τη δέσμη μέτρων και ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του σε αυτό το σημείο. Ως ε, ανέφερε και ο πρόεδρος Αρτουή, Έχουμε και κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν το 2015 γιατί η κατάσταση επήγει. Οπότε και εμεί θα πρέπει να λάβουμε το συντομότερο κάποια μέτρα. Και την Τετάρτη έχουμε την πρόταση Κομισιόν για αύξηση των πιστώσεων ε, ε, για το ΑΜΙΦ για τις ε, τρεις μονάδες των συνόρων το, το, όργανο χούντ και αυτό θα είναι της τάξης των 300 και κάτι εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει μία δεσμή μέτρων που να είναι κάτι το χωριστό από τα όσα διαπραγματευόμαστε για το σχέδιο του 16. Να καλύψουμε δύο χρόνια. Αλλά το σχέδιο τροποποιητικού προπολογισμού του 2015 θα μπορούσε να προχωρήσει με συνεννόηση των δύο θεσμών οργάνων και να εγκριθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, ούτω ώστε να εκταμιευθούν τα χρήματα προ εκείνου που τα χρειάζονται το συντομότερο δυνατόν. Και αυτό να μην καλυφθεί από την διαδικασία συνεννόησης για το σχέδιο προπολογισμού της χρήσης του 16 και τον Μάιο. Αυτό το οποίο προτείναμε θεωρήσαμε ότι είναι υπεύθυνο σχέδιο προπολογισμού, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και το σχέδιο των πληρωμών. Από τότε δε συμφωνήσαμε όσον αφορά ε, το ΕΨΙ για στρατηγικές επενδύσεις και επίσης είπαμε ότι θα καλύψουν τον προπολογισμό, τις προκλήσεις αλλά και αυτές τις κρίσεις. Αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνη αντιμετώπιση. Μια που δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο για το 3, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται την ευελιξία που χρειάζεται το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και επίσης να τηρήσουμε την δημοσιονομική πειθαρχία που απαιτεί το κάθε ευρώ να αποδίδει. Ακριβώς όπως ε, είπαμε για τα θέματα υψής της προτεραιότητας για το Κοινοβούλιο. Και τώρα, με λίγα λόγια, να σχολιάσω τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Και με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι έχουμε ένα σώρο τροπολογίες του Κοινοβουλίου που είναι συνολικά τροπολογίες 1270 όπως είπε και ο πρόεδρος και σε μεγάλο βαθμό ε, τηρούνται τα όσα δεσμευτήκαμε να κάνουμε για στο σχέδιο προϋπολογισμού το δικό μας για το 2016 και έτσι ανετράπησαν οι περικοπές που είχε προτείνει το Συμβούλιο. Σε κάποιες περιπτώσεις πάντως το Κοινοβούλιο προτείνει σημαντικές αυξήσεις πέραν του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016 της Κομισιόν. Να σας πω με δύο λόγια ποιες είναι αυτές πρώτα-πρώτα όσον αφορά το κονδύλιο 1α είπαμε ότι κάποιες πολιτικές ομάδες και κάποιες επιτροπές θέλουν να επανέλθει ε, η πίστοση υποχρέωση για το 2020 και το Connecting Europe Facility. Ακριβώς όπως είχε και πριν έχουμε το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων. Ε, να μην ε, επιμείνουμε όσον αφορά τη δική μας γνώμη για αυτά τα οποία λέει ο κύριος ε, Φερνάντες και με τον οποίο συμφωνούμε, δηλαδή απασχόληση, επιχειρήσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί μια που ε, στο, στο κονδύλι 1α δεν έχουμε μεγάλη ευελιξία και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ε, όργανο ευελιξίας για τους μετανάστες στο κονδύλι 3ε. Οπότε θα πρέπει ε, οι λίγοι πόροι που υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τι προτεραιότητες. Τώρα για το κονδύλιο 1β έχουμε διάφορε τροπολογίε. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να καλύψουμε την πρωτοβουλία για τους νέους. Να υπάρξει παράταση του σχετικού προγράμματος, Αλλά κατά τη γνώμη μας θα ήταν πρόημο να έχουμε τώρα δεσμεύσει ε, κονδυλίων από τώρα γιατί τα προγράμματα θα συνεχίσουν να τρέχουν μέχρι το 2018 και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται επί τόπου και έχουμε ε, front loading αλλά και προχρηματοδότηση ενός δις όπως θα θυμάστε. Οπότε αυτά έχουν εκταμιευθεί πλήρως και πληρωθεί. Οπότε ο βαθμός ε, απορρόφησης και εφαρμογής θα προχωρήσει 2016-2018 Επομένως θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και επομένως να μην βιαστούμε να έχουμε δεσμεύσεις κονδυλίων για τον προϋπολογισμό του 2016. Και τώρα να κλείσω λέγοντάς σας ότι συμφωνούμε ότι θα πρέπει οι πληρωμές να ξαναγυρίσουν όπως έχουμε προτείνει εμείς, να διορθώσουμε τα όσα προτείνει ω περικοπές το Συμβούλιο, όλα αυτά να τα συζητήσουμε εις βάθος στις 19 Δεκάτου που θα συνηθούμε για τις πληρωμές. Επίσης να σας πω το πόσο συμφωνούμε με τόσο προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή Φερνάντε που θέλει για τις διοικητικές δράσεις να επανέλθουν οι προτάσεις και για τις κεντρικές ε, υπηρεσίες συμφωνούμε με όσο προτείνεται αλλά όσον αφορά τους τομείς όπου έχουμε νέες προτεραιότητες και νέες αρμοδιότητες αυτών των αποκεντρωμένων ε, ε, υπηρεσιών, όπως ας πούμε για την περίπτωση των υπηρεσιών των, με, των ε, υπηρεσιών για τη μετανάστευση, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το 5% περιοχή που είχε προταθεί. Έχουμε τη Frontex, την Άσο, την Europol, όλε αυτέ τι υπηρεσίε. Και για αυτέ τι υπηρεσίε πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτέ να ενισχυθούν οι υπηρεσίε. Δεν θα πρέπει να καλυφθούν από το όριο εκείνο του 5% και σε λίγες εβδομάδες πρόκειται την επιστολή εκτελεστότητα θα σας την ε, διαβιβάσουμε οπότε αυτό θα αφορά και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και περιμένω πώς και πώς να τα πούμε την Τετάρτη που θα έχουμε και την Αντιπρόεδρο Γεωργίευα εδώ. Οπότε τότε θα έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το σχέδιο διευθυντικού προπολογισμού. Κάτι γνώμη μας, αυτό θα είναι παράδειγμα προς για το πώς μπορούν να συνοηθούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ταχαίως να βρίσκουν λύσεις για τόσο πιεστικά προβλήματα όπως το μεταναστευτικό. Merci, euh, Σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας, κυρία εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι χάρηκαν για τα συγχαρητήρια που δώσατε οι εισηγητές. και στην ψήφο μας ε, στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια και μετά από αυτά δηλαδή η συνδιαλλαγή θα είναι βέβαια σημαντική στιγμή και λόγω και του κειμενόμενου χαρακτήρα της καταστάσεως ίσως θα χρειαστεί ακόμη να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Όπως και αν έχουν τα πράγματα θα χρειαστεί να βρούμε και ταχαίως μάλιστα λύσεις γιατί θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την κρίση του μεταναστευτικού που μας καλεί να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και χωρίς καθυστέρηση. Και για το 5% μείωση του δυναμικού των οργανισμών θα, θα απαιτήσει και αυτό μια απόφαση που είναι δίκαιη κατά τη γνώμη μου. Ο κ. Μπέγκε, νομίζω. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα καθυστερήσω ίσως με την παρέμβασή μου λίγο την διαδικασία. Τα όσα εξήγησε μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συζητηθούν εντατικά μάλιστα και σε συνδυασμό και με όσες προτάσεις θα κάνει ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να με συμπαθάτε όμως, απευθύνομαι στην εκπρόσωπο, Εάν πρόκειται να δείξουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι σε θέση να δράσουν ταχαίω, τότε για κοιτάξτε λίγο την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξέδωσε την προηγουμένη εβδομάδα. Οι χώρε μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώ ακολουθούν το παράδειγμα του Σαλιγκαριού. Να σα εξηγήσω γιατί. Λέτε και δικαίω ότι η κατάσταση του παγκόσμιου προγράμματο προγράμματος διατροφής είναι τέτοια που παρακαλούνται οι χώρες μέλη να αποδεσμεύσουν το δυνατόν συντομότερο τα κονδύλια του 2014. Και στον πίνακα που μπορείτε ακόμη να βρείτε, ο μέσος όρος των χωρών μελών, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά είναι νούμερα του τέλους του Σεπτεμβρίου, δεν έχουν φτάσει καθόλου τα κονδύλια εκείνα για το Παγκόσμιο πρόγραμμα διατροφής που θα έπρεπε να έχουν φτάσει. Και αν εξετάσετε προσεκτικότερα, στα τέλη του έτους βεβαίω είναι γνωστό ότι αυξάνεται η αποδέσμευση κονδυλίων προς τα τέλη του έτους. Ένα όμως από ένα μέρος της δραματικότητας αυτής της κατάστασης των προσφύγων οφείλεται και στο ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά στα ίδια τα στρατόπεδα προσφύγων διότι τα διεθνή προγράμματα δεν έχουν πλέον τα κονδύλια για να μπορέσουν να χειριστούν κάπως επιτυχώς την κατάσταση των ανθρώπων αυτών τόπου, εκεί όπου βρίσκονται τώρα. Άρα δεν πρόκειται μόνο για έκκληση προς τις χώρες μέλη αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι σε σύγκριση με τα νούμερα του 2014 περί τα μέσα έως τέλη Σεπτεμβρίου βλέπουμε ότι από τα κονδύλια αυτά δόθηκαν 47% λιγότερα από ό,τι τα κονδύλια του προηγούμενου έτους. Και βεβαίω δεν συγκρίνονται τα νούμερα μεταξύ των ετών, διότι η δραματικότητα της καταστάσεως έχει αυξηθεί εκθετικά. Διαπιστώνω ότι προφανώς και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μέσα στις διαδικασίες μας δεν διαθέτουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς για να μπορούμε να αντιδρούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κρίσεις. Όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία του προπολογισμού, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολήσει συλλογικά πολύ εντατικά. Το ίδιο ισχύει για την διαπίστωση, όπου πάλι γράφετε εσεί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ότι συνολικά λείπουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της ανθρωπιστικής βοήθειας για την κρίση στη Συρία για το 2015. Και προτείνεται τώρα οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουν τουλάχιστον την δέσμευση να αποδεσμεύσουν τουλάχιστον το μισό του ποσού αυτού. Μιλούμε όμως για ποσά του 2015, χωρίς να έχουμε συζητήσει καθόλου για τις ανάγκες του 2016. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να απευθύνω έκκληση επιτέλους να σοβαρευτείτε. Να σοβαρευτείτε και βλέπω ότι αυτά τα πράγματα έρχονται σε αντίφαση με τα όσα δήλωσε το Συμβούλιο των Υπουργών που δήλωσε ότι για το World Food Program θα διαθέσει τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Προχωρήστε, κάντε κάτι ταχύτατα σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Υπουργών, ακολουθήστε μια διαδικασία fast track, γιατί έρχεται ο χειμώνας Ο πρόεδρος κ. Σαρατουή. ευχαριστώ για τις υπενθυμίσεις σας και για τον κόδωνα συναγερμού που κρούεται. Η κυρία Γεωργίευα θα έλθει την Τετάρτη, περί τα τέλη του πρωινού ή αρχές του απογεύματος. Θεωρώ ότι τότε είναι δυνατόν να διεξαχθεί συζήτηση για την κρίση του μεταναστευτικού και να επανέλθουμε τότε στους αριθμούς που αναφέρατε πριν από λίγο διότι αν δεν δοθεί απάντηση και μάλιστα αμελητή στις ανάγκες των στρατοπέδων αυτών στην Τουρκία, στην ε, Ιορδανία, στον Λίβανο, τότε η ίδια η Ευρώπη θα πληγεί. Δεν είναι μοιραία τα κύματα των προσφύγων. Ελπίζω ότι και οι αρχοί κρατών και κυβερνήσεων θα συναγάγουν τα συμπεράσματά τους από την κατάσταση αυτή και θα ξεφύγουν πια από αυτή την θέση ακινησίας που οδηγεί σε απόγνωση τους πολίτες. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε τώρα, μπορούμε τώρα μάλλον να περάσουμε στην ψηφοφορία. Και χωρίς αμφιβολία θα υπάρχουν και επαληθεύσεις, δηλαδή ηλεκτρονικές επαληθεύσεις με ονομαστική ψηφοφορία. Και γι' αυτό προτείνω να κάνουμε πρώτα ένα τεστ, να βάλετε δηλαδή όλοι και όλες τις κάρτες σας στην σχισμή που βρίσκεται στο έδρανό σας, να διεξαγάγουμε μια ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Δεν έχει κανένας πρόβλημα με την λειτουργία της κάρτας. Α, η ψήφος μου περισσεύει. Μην ε, εκπλαγείτε λοιπόν, δεν θα ψηφίζω. Άλλωστε είμαι και υποχρεώμαι κιόλα να παραμείνω ουδέτερος. Θα ψήφισα μόνον εάν δεν εξαντλούσε την ποσοστοσή της η ομάδα μου. 35 λοιπόν ψηφίσαντες. Δεν φαίνεται το μηχάνημα να έχει κανένα πρόβλημα. Ας έλθουμε τώρα στο τμήμα 3 τις διοικητικές δαπάνες. Και θα ήθελα να σας δηλώσω ότι πρέπει να τοποθετηθούμε επί συμβιβασμών, συμβαστικών τροπολογιών, που είναι αυτές που πρώτες θα τεθούν όλες μαζί σε ψηφοφορία. Έχουν ζητηθεί ε, ψηφοφορίες για ορισμένες τροπολογίες και με την σύμφωνη γνώμη σας θα αρχίσουμε από τις συμβαστικές τροπολογίες. Μετά θα προχωρήσω σε ψηφοφορίες χωριστά για τροπολογίες που έχουν ζητηθεί να ψηφιστούν και εάν βέβαια ε, υπερψηφιστούν αυτές υπερισχύουν των όσων έχουν ενταχθεί στους συμβασμούς. Πρώτος συμβασμός λοιπόν, τμήμα 3. Κονδύλια 1 έως 4, διοικητικές δαπάνες, ψήφι υπέρ του συμβασμού αυτού. Ποιο λέει ρε παιδιά. Τώρα, ποιο λέει ρε παιδιά. Abstention. Κατά αποχές, αυτός ο συμβασμός εγκρίνεται. Δεύτερο μπλοκ 5-3 δαπάνε, θέτω σε ψηφοφορία ψήφι υπέρ Σας ευχαριστώ. Αποχέ, εγκρίνεται και ο δεύτερος αυτός συμβασμός. Τώρα, ψηφοφορίες χωριστές. Μια πρώτη τροπολογία της κυρίας Γκρέσλε, α30301, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Χιχι μέχρι 11 0-1 βάλουμε 2-11 ψήφι υπέρ κατά θα κάνουμε παρήθεση με ηλεκτρονική ψηφοφορία Le scrutin est clos. Pérasse. Εγκρίνεται η τροπολογία αυτή με ψήφους 19 υπέρ, 16 κατά. Ο κ. Σάρβαμα 10-01-05-15. Α, πρώτα υπάρχει μια συμβαστική τροπολογία που καλύπτει 70 και η τροπολογία Σάρβαμα 4.360. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής αυτής της τροπολογίας. Ευχαριστώ. Αντίθετη. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, η επόμενη τότε εκπίπτει αφού εγκρίθηκε η συμβαστική, η 32.01.05.21, τροπολογία Ήτρε 52.90, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32-01-05-23 52-91 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 21-01-04-04 τροπολογία Φεραίρα της Επιτροπής Υπολογισμών υπέρ κατά αποχές αυτή απορρίπτεται. Περνούμε στα σχόλια και ονοματολογία. Στο 29.01.04.01 τροπολογία Φερέιρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Στην 19.01.04.01 Γονζάλες Πένιας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16.03.02.04 Τροπολογία Μούντι Χόιτ υπέρ. Κατά να προχωρήσουμε σε επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει. Τέλος. Απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Στην 3.01.01 ε, S0202 Γκρέσλε υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται αυτή στην 31.01.07.01 τροπολογία Ζούμπερ υπέρ κατά αποχές αυτή απορρίπτεται στην Χ01 τροπολογία 74.13 της Ενωτικής Αριστεράς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυτή αποθεματικά 32 01 05 23 η 77 40 των πρασίνων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην 30 01 13 01 της κυρίας Κρέσλη 43-10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24-01-07 και α3-01-01-01 τροπολογία Κρέσλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή Τελείωσε, τελείωσαν μάλλον οι διοικητικέ δαπάνε του τρίτου τμήματος. Και περνάμε στις, στους οργανισμούς. Για τους οργανισμούς αρχίζουμε όπως και προηγουμένως από τις συμβαστικές ε, τροπολογίες τα μπλοκ και μετά θα περάσουμε στις ε, μεμονωμένες τροπολογίες. Η πρώτη δέσμη τροπολογιών, το πρώτο μπλοκ, επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική πρόταση. Δεύτερο μπλοκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και η δεύτερη δέσμη. Τρίτη δέσμη. Υπέρ. Κατά. Δεν είδα να σηκώνονται όλα τα χέρια. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και τρίτη δέσμη συμβαστικών τροπολογιών και περνάμε στις μεμονωμένες τροπολογίες γραμμή 180203 και 1802030102 για τη Frontex. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτεται με 15 ψήφους υπέρ και 18 κατά. Δύο αποχές. 17.03.10 Τροπολογία 46.20 Ποιος είναι υπέρ, κατά Αποχές Απορρίπτεται 18.02.03 82.00 των μεταρρυθμιστών συντηρητικών ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18.02.04 μεταρρυθμιστή συντηρητική 82.07 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33.02.07 ECR 82.06 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στα αποθεματικά. 12.02.06. Τροπολογία Giggold 44.95. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στις παρατηρήσεις ε, γραμμή 040311 Επιτροπή Γυναικών 6009 ε, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 040312 Επιτροπή Γυναικών 625. ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 4002 καλύπτεται 06-02-03-02 Τροπολογία Επιτροπής Προϋπολογισμών 41-36 του κ. Νεγκρέσκου. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12-02-05 Τροπολογία της Επιτροπής ΕΚΟΝ 63-09. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Άποχες εγκρινεται 7538 τροπολογία του ΕΛΚ καλύπτεται. Το ίδιο και των σοσιαλιστών, 70-39. Τροπολογία φιλελευθέρων, 80-02. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41-05 της Επιτροπής Προϋπολογισμού του κ. Άλλη. Καλύπτεται από την προηγούμενη. Δεν θα ψηφίσουμε. 32.02.10 53.04 τη Ήτρε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18.02.03 Τον πράσινο ποιος είναι υπέρ. 77.18. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18.03.02 της ΛΥΜΠΕ 59.98 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή των γυναικων 60.21. για την τροπολογία για την γραμμή 18.03.02 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4631 των προϋπολογισμών καλύπτεται. Γραμμή 330207 της Επιτροπής Γυναικών η τροπολογία 633 καλύπτεται και αυτή από την πρώτη συμβαστική δέσμη. Οπότε ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες ε, για τους οργανισμούς και περνάμε στο τμήμα 1α Heading 1α. Ίδια διαδικασία με αυτή που ακολουθήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή πρώτα θα δούμε τις συμβαστικές τροπολογίες που είναι δέσμες συμβαστικών τροπολογιών και κατόπιν θα εξετάσουμε τις μεμονωμένες τροπολογίες. Πρώτο μπλοκ που ζητά επαναφορά των πιστώσεων του σχεδίου προπολογισμού. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, δεύτερη υποκατηγορία συμβαστικών τροπολογιών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτη δέσμη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Περνάμε τώρα τις, στις μεμονωμένες τροπολογίες. Καταρχήν, δημοσιονομική γραμμή 010104. Έχουμε δύο τροπολογίες, μία της ΓΚΟΕ την 7415 και τον προϋπολογισμό 4389. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Γραμμή 010201. Τρεις τροπολογίες, πανομοιότυπες, η FDD 7850, GUE 5 και η προπολογισμό 4390. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Γραμμή 010406. Η FTD 7851. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 02-02-02 γκουε 72-64 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται γραμμή 02-04-02-03 γκουε 72-67 ποιος είναι υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Έχουμε δύο πανομοιότυπες τροπολογίες ε, για τη 04-0265 και 04-07. Γκου 74-14, προϋπολογισμοί 44-23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Γραμμή 04-03-01-01. Γκου 72-74 και ε, ποιος είναι υπέρ μάλλον. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία της ΕΣΥΑΡΙ 8202. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 04-03-01-05 ECR 82-04. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 04, 03, 01, 06 EFDD 7866 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 04, 03, 01, 08 EFDD 7853 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 04, 03, 02, 01. ECR 82, 05. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 06, 02, 05. Η FTD 78, 78. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12, 02, 01 δύο τροπολογίε ταυτόσημες, η FDD 7888 και προυπολογισμοι 4451. 44-51. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. 140401. Απορρίπτονται. 4609. προυπολογισμοι Προϋπολογισμοί είναι υπέρ? Κατά. απορριπτεται 150202. επιτροπη προπολογισμών 4615. 46-15. είναι υπέρ? κατά αποχές απορρίπτεται. Αποθεματικά τώρα. Για τη γραμμή 120203. Τροπολογία σοσιαλιστών, 7148. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία ΕΚΟΝ 6305. Καταπίπτει μια και εγκρίθηκε η προηγούμενη των σοσιαλιστών 48. Η μοίρα έχει και η τροπολογία 4494 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Τροπολογία 3205-0101. Τροπολογία 41.11 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Αποσύρεται η τροπολογία για την 3205-0102. Τροπολογία των Πρασίνων 77.41. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41-12 της Επιτροπής Προϋπολογισμών αποσύρεται παρατηρήσεις. Για τη δημοσιονομική γραμμή μηδέν 4390 της Επιτροπής Προϋπολογισμών αλλά καλύπτεται από τις συμβαστικές τροπολογίες απορρίφθηκε 02-01-06-01 41-33 της Επιτροπής Προϋπολογισμών ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 02-02-01 πρώτη τροπολογία 43-98 της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Μπάτς Ψηφοφορία κατά τμήματα. Για το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. Δεύτερο τμήμα αποσύρεται. Δύο τροπολογίε φιλελευθέρων, 8079 και badge 4107. Πανομοιότυπε οι τροπολογίε με νέα διατύπωση. Δεν χρειάζεται να στη διαβάσω. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 60.00 της Επιτροπής Γυναικών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, Γκουε. 72.61 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπάτζ 4393. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκόν 6323. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για τη δημοσιονομική γραμμή 020202, τροπολογία ΚΟΕ 7263, με νέα διατύπωση. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ, με ονομαστική κλίση θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, γιατί δεν είδα είναι ψηλά όλα τα χέρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22 ψήφοι κατά, 13 υπέρ. Μπατ 4399, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φαμ 6001, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 ψηφιπέρ και 18 κατά. Δύο οι αποχές. Στην δημοσιονομική γραμμή 020301, τροπολογία badge 4061, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40-64 της Μπάτς. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στη δημοσιονομική γραμμή 02-03-02-01 έχουμε την τροπολογία ΦΑΜ 60-02. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Mm. Για τη 0204, τροπολογία ΦΑΜ 6003, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γραμμή 0204-0202, τροπολογία 6004 ΦΑΜ, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για τη γραμμή 0203 τροπολογία ΦΑΜ 6005, Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 15 ψηφί υπέρ, 18 κατά. Δύο αποχές. Δημοσιονομική γραμμή 02, 04, 03, 01. Μπατ 41, 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 04, 03, 01, 03. Δύο τροπολογίες ταυτόσιμες των σοσιαλιστών 70-45 και μπατ 40-85. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Για την ίδια γραμμή τροπολογία ΦΑΜ 6007. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία της Επιτροπής Απασχόλησης 6260. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Στη δημοσιονομική γραμμή τροπολογια μπατση 4140. 41-40. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4266. 42-66. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Για τη 04, 03, 01, 05, τροπολογία μπάτ 41, 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, η FAM 6024 και BADGE 4001, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 18 ψήφοι κατά, 15 υπέρ, 2 αποχές. Για τη γραμμή 04-03-01-06, Επιτροπή Απασχόληση, Τροπολογία 62-97, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Για τη 04, 03, 02, 01, τροπολογία μπάτσα 42, 62, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Για τη 04, 03, 02, 03, μπάτς 41, 35, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επιχειρηματικότητα. Τροπολογία 6208 της Επιτροπής Απασχόλησης. Με προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία της Επιτροπής ΦΑΜ. 6008. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για τη γραμμή 06020101, τροπολογία των Πρασίνων, 7722, ε, την έχουν αποσύρει. Στη γραμμή 06-02-01-02, Επιτροπή Transport Μεταφορών 56-11, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για τη γραμμή 08 έχουμε την τροπολογία badge 40-70, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία ε, φάμε 60-10. Ποιος είναι υπέρ για τη γραμμή 08-02-01. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται. 08-02-02-02. Τροπολογία φάμε 60-11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 08-02-02-03 μπατ 42-38 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γραμμή 09-03-02 μπατ 41-38 ποιος είναι υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται στη γραμμή 14-03-01 τροπολογία 41-42 της Επιτροπής Προπολογισμών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται γραμμή Batch 41-46. ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Γραμμή 15-02-01-01. Τροπολογία φιλελευθέρων. 80-27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται στην ίδια γραμμή η τροπολογία 612 της ΦΑΜ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γραμμή 150203 Επιτροπή Πολιτισμού 5812 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Γραμμή 1503. Επιτροπή Γυναικών 6013. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γραμμή 240201. Μπάτς 4143. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 290201. Μπάτς 4586. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40-50 της Επιτροπής Προπολογισμών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ήταν η γραμμή 32-02-01-02. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 32-02-02. Μπατ 40-51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και ολοκληρώσαμε το 1α. Περνάμε στην κατηγορία 1β μικρό. Και ευθύς αμέσως αρχίζουμε τις ε, πιο χωρισμένες ψηφοφορίες. Γραμμή 040260. Έχουμε μια τροπολογία, δύο διόρθωνα προϊόντα, δύο ταυτόσιμες τροπολογίες. Αποσχόληση 62-43 και των πρασίνων 77-28. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται 04-02-61 των πρασίνων 77-30. Και ΕΟΥΡ ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρασινών. 77-31. Και ΕΟΡ 2-3-8-14-54. που είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 04-02-62. Απασχόλησεως 62-04. έω 2 εκατομμύρια. Ευρώ δηλαδή. που είναι υπέρ, που είναι κατά. Αποχές απορρίπτονται. 64 Πρωτοβουλία για τους νέους. Πρώτα πρώτα έχουμε μια συμβαστική τροπολογία ε, του εισηγητή υπέρ της συμβαστικής. Κατεβάσα τα χέρια. Κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική. Επομένως, ε, οι επομένες ε, τροπολογίες για την ε, ίδια γραμμή Κατά καταπίπτουν. Και πάμε στο 0406-01. Επιτροπή. Προπολογισμό 44-47. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 62-31 της Ευρωπασχόλησης και 20 εκατομμύρια υπέρ, κατά, αποχές Απολύτωται. η υπομένη αποσύρεται 040602 6293 της απασχολήσεως και ταυτόσημη της 44-12 προϋπολογισμών και ευρώ 1 εκατομμύριο 60.000 ευρώ υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 13.03.63 της ΓΚΟΥ 73.01 προϋπολογισμών 43.24 ευρώ 6 εκατομμύρια και κάτι υπέρ κατά αποχές απορρίπτωτο 13.04.60 Γκουε 73.02 προϋπολογισμοί 46.06.18 εκατομμύρια και κάτι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22.04.03.02 άφετ 50.35 6 εκατομμύρια και κάτι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Αποθεματικά 13.03.60 Τροπολογία Γκρέσλε 43.06 Πέρα κατά αποχές απορρίπτεται 13.03.62 προϋπολογισμοί 43.07 Γκρέσλε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13.04.60 40.63 προϋπολογισμών Μπέλτερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Και τώρα, οι υποσημειώσει παρατηρήσει 040260, προπολογισμοί 4062 Μπέλτερ, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 040264, γκου 7273, 4407 προπολογισμοί υπέρ. Κατά. Αποχέ θα πρέπει να γίνει έλεγχος ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτωται. 23, 11, μία εποχή. Συνεχίζουμε. Γυναικών, 60, 06, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίδια γραμμή, προπολογισμοί 42-47 μπέγγι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογισμοί 42-65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. 04-06-01. Προπολογισμοί 44-47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 06, 02, 01, 04. Πράσινη, 77, 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Προϋπολογισμοί Προϋπολογισμοί 06 Γκρέσλε υπέρ Κατά Αποχές Απορρίπτωται. 13-03-62. Προπολογισμή 43-07 γκρέσλε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 13-03-63 γκου 73-01 προπολογισμή 43-24. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 13 03 Σοσιαλιστές και Δημοκράτες 70-48 υπέρ κατά Αποχές Απορρίπτεται 13-04-60 Γκουε 73-02 Υπέρ Κατά Αποχές Απορρίπτεται Για την ίδια γραμμή προϋπολογισμή 46-06 Υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Nous με την κατηγορία 1β. Πάμε τώρα στο κονδύλι 2. Και σύμφωνα με την ε, διαδικασία, όπως έχει αυτή συμφωνηθεί, θα ψηφίσουμε τις δύο ομάδες τροπολογιών κατόπιν ε, συμβιβασμού. Η πρώτη υποδέσμη, οπότε και επανέρχονται τόσο να συμφωνηθεί για το σχέδιο προπολογισμού. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται αυτή η δέσμη τροπολογιών, δεύτερη τώρα, υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε τις καθέκας των τροπολογίες. 05-02-03 πράσινη. Αφού 10 υπέρ. Κατά. Θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Le scrutin est clos. Πέρασε. Απορρίπτεται Γκουε 72-85 Υπέρ Κατά Αποχές Απορρίπτεται. 05-02-08 12 προϋπολογισμοί 44-30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται την διαγραμμή 70-32 σοσιαλιστές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 05-02-12-08 Σοσιαλδημοκράτες 70-33 υπέρ κατά Είμαστε και ψηφοφορία. ψηφίζουν πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 20, 11, 2 εποχές. 05, 02, 13, 01, πράσινη, 77, 08, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 05, 03, 11. Προϋπολογισμοί. 43, 61, σορβαμά, υπέρ. Qui s'abstient L'amendement est repoussé. Απορρίπτεται η τροπολογία. 05, 08, 80, πράσινη 77, 16. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 07, 01, 04, 01. Γκου 72, 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11, 03, 03. Γκου 72, 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Φερέιρα. Επίσης απορρίπτεται. 11.73.03. Γκου 72.99 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Γραμμή. 11.0660. Τροπολογία Γκου. 72.98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11.0662 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11.0665 Τροπολογία 44.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αποθεματικά 05, 03, 01, 10 44-93 προϋπολογισμοί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα υποσημειώσεις παρατηρήσεις 05-02-05-99 Γεωργία 54-23 υπέρ κατά αποχές απορριπτεται 05 05-02, 502-12-99. 54-26 Γεωργία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμοί. 40-41 είναι ταυτόσιμοι. Άρα και αυτή ακολουθεί την τύχη της προηγουμένης. 05-03-01-01. Περιβάλλον 61-44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 05-03-01-10. Προϋπολογισμοί 44-93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η διαγραμμή. Πράσινη 77-12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 07, 02, 01. Σοσιαλδημοκράτες. 70, 47. Α, καλύπτεται από την συμβιβαστική. C'est Καλύπτεται όπως καλύπτεται και η επόμενη. Άρα πάμε στο 07, 02. Α, ευχαριστεί το λόγο κύριο Σταράν. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά θεώρησα ότι εγκρίθηκε η τροπολογία που αφορά τις ε, ταυρομαχίες, ε, τις θανάσιμες, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Για να το κοιτάξουμε τώρα. Le, le, votre amendement a été repoussé. η τροπολογία που εννοείται. Θέλει να γίνει έλεγχος. Ναι, λέει ο βουλευτής. Όχι, λέει. Απερίφθηκε. Pardon Alors un contrôle. Ωραία, θα γίνει έλεγχο. Ψηφίζουμε. Ποια ψηφίζουμε? Την 77-12. Ε, 77-12. Να μην υπάρχει ενίσχυση των θανάσιμων ε, ταυρομαχίων. Πέρας. Α, il est adopté. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 16-15 και τρεις αποχές. Je vous demande pardon, mais moi je n'avais pas vu. Bien, on a dit que. Το 070201 καλύπτεται από την συμβαστική. Το 070202 ε, και η προπολογισμό 4059 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτη τροπολογία. 6703. 5425 Γεωργία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ο κύριος Σαρβαμά όμως θέλει να γίνει έλεγχος για το 44-93 στην ίδια σελίδα. Οπότε θα κάνουμε έλεγχο για την Μητροπολία Σαρβαμά. 44-93 προϋπολογισμών. 05, 03, 01, 10 ήταν η, η τροπολογία. 05, 03, 01, 10. Ligne 05-03-01-10 05-03-01-10 44-93 προϋπολογισμών Le scrutin est Ψηφίζουμε. Oui, oui, bah, c'était Πέρασε. Απορρίπτεται η τροπολογία. 20-15. Αφού θέλετε έλεγχο, να το ζητείτε ευθύ αμέσω την ανακοίνωση του αποτελέσματο τη ψηφορία. Ολοκληρώσαμε εδώ γιατί το 42 προϋπολογισμών, 40-42 συγγνώμη, είναι ταυτόσιμο με την προηγούμενη τροπολογία, η οποία απερίφθη. Οπότε ολοκληρώσαμε και με την κατηγορία 2. Euh, Sur la rubrique 3. Κατηγορία 3. Συνεχίζουμε. Εξήμιση οφείλουμε να ολοκληρώσουμε. Αν δεν έχετε πρόβλημα, να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε την κατηγορία παριθμών 3. Έχουμε εδώ τρεις δέσμευσες ε, τροπολογιών όπως προέκυψε από τους συνδεσμούς. Πρώτον, ψηφίζουμε. Είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη δέσμη τροπολογιών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτη δέσμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα οι καθέκες των τροπολογίες που δεν καλύπτονται από αυτές τις δέσμες τροπολογιών κατόπιν του συμβασμού 17.04.01 προϋπολογισμή 24 υπέρ κατά αποχές απολύπτεται περιβάλλον 61.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γραμμή 18-01-06-01 προπολογισμή 45-02 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 18-02-01-01 προπολογισμή 45-01 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18-02-01-02 προπολογισμή 44-91 υπέρ. Κατά αποχες απορριπτωτα 18 απορρίπτεται 18-02-01-03-46-27 προϋπολογισμοί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18-02-01-04-73-18 γκουε προϋπολογισμοί 44-96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18.02.08 προπολογισμή 43.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18.03.03 προπολογισμή 46.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18.02.01.04. Έχουμε μια τροπολογία σοσιαλδημοκρατών 7046. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 22-11 2 εποχές. Και τώρα για τις πιστώσεις αμύφ. 18-03-01-01-02-03-04 και 05. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Europe for Citizens πρωτοβουλία. 18.04.01.01 και 02. Αύκο 65.60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επομένη. Καταπίπτει. Παρατηρήσεις, υποσημειώσεις 09.05.05 πολιτισμού 58.07 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15.04.01 απολυσμό 58.43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16.03.01.02 αυκό 65.50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16.03.04 προϋπολογισμοί 30.40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17.03.01 Αλντέ 875 Συν προφορική του εισηγητού. Έχετε το κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17.04.01 41.48 προπολογισμό. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Απορρίπτονται. 17.04.02 Γκου 73.25 προπολογισμή 46.25 Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 17.04.04. Ε, 17.04.03 προπολογισμό 40.60 υπέρ κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά ας κάνουμε επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται 18-17 17-04-04 Γκούθινα 3-27 Προπολογισμή 6, Ταυτόσημη Ταυτόσημης υπέρ κατά Αποχές Απορρίπτεται Γραμμή 18-02-01-01 γυναικών 60-14 υπέρ κατά επαλήθευση ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 22 11 δύο εποχές Για την ίδια γραμμή, δύο τροπολογίες ταυτόσιμες, γκουε, 73-16, προϋπολογισμοί, 45-0-0, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτονται. Απορρίπτονται. Σωστό το λέει ο 18-02-01-02. πρώτον 97 προϋπολογισμοί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμών. 40-57 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 20-14 με μία εποχή. Στην ίδια γραμμή της Γκουερ. 73, 17. Υπέρ, κατά. Αποχής. Απορρίπτεται. Ίδια γραμμή. Προϋπολογισμό 44, 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 01. Γυναικών 641 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Η 73-19 της ΓΟΕ και τον προπολογισμό 43-31, οι οποίες είναι ταυτόσιμες, τις ψηφίζουμε τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτονται. 18-03-01-02 προπολογισμο 45-04 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. 18.04.01 προϋπολογισμών 41.15 με μια προφορική τροπολογία έχετε το κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33.02.01 προϋπολογισμών 45.97 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 60-23 γυναικών 74-07 προπολογισμό 45-96 ταυτόσιμες. Τις ψηφίζουμε όλες μαζί υπέρ κατά επαλήθευση. Ψηφίζουμε τώρα. πέρας. Απορρίπτεται 19-15. 33-02-02 γυναικών 60-42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33-03-01 γυναικών. 60-26. Προπολογισμό 40-03 ταυτόσημες ειμαι υπερ Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι. Με εντατικό ρυθμό προχωρήσαμε, οπότε μπορούμε να βάλουμε τελεία για απόψε σε αυτό το σημείο και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας αύριο το πρωί για την κατηγορία 4. Θέλει κάποιος το λόγο? Ουδής. Άρα θα συνεχίσουμε αύριο στις ε, μισή. Όχι, 9, 9. 9 διορθώνει ο πρόεδρος. Εδώ. bon, l'observation.